Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο διορισμός σας είναι ιστορικός. Είσαστε ο πρώτος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχει αυτή τη θέση και οι δύο μας οργανισμοί προέκυψαν από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προωθώντας την ειρήνη και την ευημερία μέσα στα πλαίσια μιας πολυμερούς συνεργασίας. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να τους δώσουμε απτά αποτελέσματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διεθνείς προκλήσεις, την ριζοσπαστικοποίηση, την τρομοκρατία, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, την φτώχεια και την ανεργία. Οι πολίτες μας περιμένουν μια Ευρώπη πιο παρούσα και αποτελεσματική στο διεθνές σκηνικό. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτωχοι στους βομβαρδισμούς της Συρίας και στον λοιμό της Αφρικής, καθώς και στο δουλεμπόριο γυναικών και παιδιών και στις μεταναστευτικές ροές καθώς και την οπισθοχώρηση της δημοκρατίας σε ορισμένες χώρες όπως τη Βενεζουέλα και την Τουρκία ή την δίωξη θρησκευτικών μειονοτήτων. Χτες μιλήσαμε για την Αφρική με τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, τον κύριο Μουσαφάτ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Αφρική είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την τριμερή συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης, Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να δώσουμε τάχιστες απαντήσεις στις κρίσεις και σειράξεις. Θα πρέπει να βρούμε κοινέ πολιτικές λύσεις για την σύραξη στη Συρία, Λιβύη και Ιεμένη και να αντιμετωπίσουμε την ΤΑΕΣ. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια και ελευθερία των ανθρώπων, να δώσουμε προοπτικές στις νέες γενναίες και να προωθήσουμε την Ατζέντα 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη. Κύριε Γενική Γραμματέα, μπορείτε να βασιστείτε για όλα αυτά στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτή την ατζέντα η οποία είναι και δική μας. Κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε το λόγο. Mr. President, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.